Τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι η έκθεση της κυρίας Μαγκίνης που έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Κύριε Επίτροπε, κύριε και πρόεδρε κυρία Επίτροπε, το πρόβλημα της έκθεσής μου ήταν όταν είχα αρχίσει να τη γράφω η προτεραιότητα, δηλαδή η επισητιστική ασφάλεια θεωρούνταν προτεραιότητα από όλους. Λόγω της κακής διατροφής που παρατηρείται παγκοσμίω. Και πολλά εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα λόγω μη επαρκούς διατροφής. Πρέπει λοιπόν να διατεθούν τρόφιμα σε όλους όσους τα χρειάζονται. Ευχαριστώ την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανάπτυξης που συμμετέσχε στο σύνολό της στην επεξεργασία της εκθεσής μου. Δεν έχω το χρόνο να σας αναφέρω όλες τις λεπτομέρειες, αλλά θα τονίσω τα κυριότερα σημεία. Πρώτον, κοινή αγροτική πολιτική και η διατροφική ασφάλεια συνδέονται προφανώς. Και γι' αυτό υπάρχει μια τάση να κατηγορούμε την ΚΑΠ για τα πάντα. Αυτό δεν είναι σωστό. Η ΚΑΠ βοήθησε τους πολίτες μας να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της διατροφής τους και ίσως να είναι και πρότυπο για το τι μπορεί να γίνει διεθνώς. Η ότι η γεωργία Βέβαια μπορούμε να πούμε ότι είχε εφαρμοστεί με λανθασμένο τρόπο τα τελευταία δέκα χρόνια. Διαπιστώσαμε δηλαδή ότι τα κονδύλια για την ανάπτυξη της υπαίθρου είχαν τύχει κακής χρησιμοποίησης. Σήμερα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο Σήμερα γίνεται λόγος για το πρότυπο που αποτέλεσε η κοινή αγροτική πολιτική και σε άλλες χώρες. Πρέπει λοιπόν σε τοπικό επίπεδο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της διατροφής και της γεωργίας και όχι με επιχορηγήσεις. Και το θέμα δεν είναι μόνο τα λοιπάσματα και οι σπόροι, αλλά και η απαραίτητη γνώση και τεχνογνωσία για να μπορέσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της διατροφής τους. Διαπιστώθηκε ότι είναι δυνατόν. Χρειάζονται βέβαια πρωτοβουλία, ανάληψη πρωτοβουλειών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει διεθνώ υπέρ του αναπτυσσομένου κόσμου πρέπει να δηλώσει προς τις χώρες αυτές ότι πρέπει να προσπαθήσουν να παραγάγουν μόνες τους τη διατροφή τους. Το πρόβλημα είναι βέβαια λεπτό. Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Κατά 40% θα αυξηθεί το 2050. Και αυτό θέτει ιδιαίτερα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα διατροφής, ζωοτροφών κλπ. Στην Ευρώπη θελήσαμε να μειώσουμε την παραγωγή τροφίμων και δεν λάβαμε υπόψη μας όλες τις δυνατότητες που είχε η δική μας γεωργία. η γεωργοί λοιπόν παράγουν όσο καιρό τους συμφέρει αυτό. Πρέπει η πολιτική να τους δίνει το κίνητρο, τη δυνατότητα μάλλον, να κερδίζουν τη ζωή τους με αξιοπρεπή τρόπο και με ανεκτό κόστος. Πριν από ένα χρόνο έγινε λόγος για τις ψηλές τιμές των τροφίμων. Σήμερα υπάρχουν πάλι πλεονάσματα και ίσως η μείωση της παραγωγής να χειροτερέψει τα πράγματα. Σας ευχαριστώ όλους και όλες πάντως γιατί δείξατε πόσο σας ενδιαφέρει το θέμα. Κυρία Βασιλείου, ευχαριστώ. Η Επιτροπή χαιρετίζει την έκθεση της κυρίας Μαγκίνες και την συζήτηση που έγινε στις διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές για το επίκαιρο αυτό θέμα που αφορά και το εμπόριο και τα βιοκαύσιμα και την παρακολούθηση των τιμών, την επενδυτική πολιτική, την αξιονομική κρίση, τις κλιματολογικές αλλαγές κλπ. Και η Επιτροπή συμμερίζεται γενικά την ανάλυση των λόγων της ε, διατροφικής κρίσης που έπληξε πολλές χώρες το 2008. Θα συνεχίσει να αναλύει την σύνδεση μεταξύ τιμών ενεργείας και τιμών των τροφίμων. Είναι πολύ το θέμα αυτό γιατί αφορά τη διασύνδεση πολλών παραγόντων ε, ζήτησης και προσφοράς. Οι ενεργειακές τιμές είναι μόνο ένας από αυτούς τους παράγοντες, αλλά υπάρχει, έχουν, έχουν οι τιμές και άμεσο και έμεσο αντίκτυπο. Το Κοινοβούλιο συζήτησε το θέμα σε βάθος και υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της πολιτικής της Ένωσης και της εν, πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν αγοράσει κανείς, αν τα βιοκαύσιμα μάλλον δεν καταλήγουν στην καλύτερη χρησιμοποίηση και των ζωοτροφών δεν καταλήγουμε πουθενά. Ακόμα και αν ο στόχος του 10% επιτευχθεί, η επίπτωση στις τιμές των τροφίμων θα είναι ελάχιστη γιατί όλο και περισσότερα βιοκαύσιμα θα κατασκευάζονται, θα παρασκευάζονται από απόβλητα. Και δεύτερον, η σοδιές τους θα συνεχίσουν να αυξάνονται και να βελτιώνονται. Μια βιώσιμη πολιτική βιοκαυσίμων της Ένωσης είναι κάτι που πρέπει ακόμη να βελτιωθεί. Οι γεωργοί πρέπει να μπορέσουν να συνεχίσουν να ζουν στην Ήπεθρο και να κερδίζουν τη ζωή τους αξιοπρεπώς. Η Κομισιόν είναι αποφασισμένη να παρακολουθήσει στενά τη σύνδεση μεταξύ ασφάλειας των τροφίμων και τιμών τους. Θέλουμε να υπάρξει σφαιρική ασφάλεια των τροφίμων μέσω της προσαρμογής στην διεθνή κατάσταση. Το λεγόμενο check-up που δεχτήκαμε πρόσθετα θα απλοποιήσει την ΚΑΠ και θα μειώσει τις, ε, τους περιορισμούς που υφίστανται οι αγρότες έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα διεθνή, τις διεθνείς προκλήσεις. Η αύξηση των ποσοστώσεων των γαλακτοκομικών πριν από την κατάργησή του το 2015 και είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει ένα πραγματικό δίκτυο ασφαλείας. Υπάρχουν και νέες προκλήσεις όπως οι κλιματολογικές αλλαγές, η διαχείριση των υδάτων, οι ανανεώσιμες πηγές ενεργείας και η βιοπικιλότηση που θα έχουν επιπτώσεις και στη ζωή των αναπτυσσομένων χωρών. Η ΚΑΠ δεν θα παραμείνει στάσιμη μέχρι το 2000, μετά το 2013 και έχουν αρχίσει οι σχετικές συζητήσεις από την πρώτη άτυπη διάσκεψη των Υπουργών Γεωργίας. Η μελλοντική ΚΑΠ πρέπει να θεωρηθεί στα πλαίσια του ανταγωνιστικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης κλπ έχουν τονιστεί δεόντως έχει τονιστεί δεόντως η σημασία που έχει η τροφιμική ασφάλεια. Υπάρχουν δεσμεύσεις και ενωσιακός και διεθνός για να τεθεί ψηλά στις προτεραιότητές μας το θέμα αυτό καθώς και της ανάπτυξης της υπαίθρου. Παραδείγματος χάρη συζητήσαμε το θέμα της γεωργίας και της τροφιμικής ασφαλείας κατά την συνάντησή μας με την Αφρικανική Ένωση τον Οκτώβριο όπου είχαμε θα και θα προσπαθήσουμε να την επαναλάβουμε τη συνάντηση αυτή. Τέλος η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθήσει τι έχουν συζητήσει οι ηγέτες του ΓΑΜΑ 8 σχετικά με την τροφιμική ασφάλεια. Στις 16 Δεκεμβρίου το Συμβούλιο συζήτησε το θέμα της τροφιμικής διευκολύνσεως και ζήτησε τη δημιουργία μιας ομάδας υψηλού επίπεδου. Η Κομισιόν προσβλέπει με αδημονία στην έγκριση του σφαιρικού πλαισίου γιατί είναι πεπισμένη ότι η γενική εταιρική σχέση σύνδεσης της γεωργίας με την τροφιμική ασφάλεια θα παίξει ρόλο κλειδί στην εφαρμογή των διαφόρων συστάσεων που γίνονται στην έκθεση αυτή μεταξύ των οποίων και πώς να προωθήσουμε τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις καθώς και το ποιες ποια εμπορικά προγράμματα είναι τα καλύτερα για να στηριχθούν οι πιο ευαίσθητες κοινότητες. Τέλος, ξέρουμε ότι ο δρόμος είναι περισσότερη απελευθέρωση του εμπορίου και όχι λιγότερη. Η Κομισιόν ελπίζει ότι το τολμηρό βήμα που έλαβαν τα, ευρωπαϊκά, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να κινητοποιήσουν ένα δισεκατομμύριο που προβλέπεται για την παρακολούθηση των τιμών των τροφίμων και βραχή και μέσο μακροπρόθεσμα θα ακολουθηθεί και από τις ανάλογες δωρεές. Η διάσκεψη της Μαδρίτης για την ασφάλεια τροφίμων για όλους στις 26-27 Ιανουαρίου σίγουρα θα αποτελέσει πολύ σημαντικό βήμα για να προχωρήσει η συζήτηση σε άλλο επίπεδο, δηλαδή στην ταύτιση των βασικών προτεραιοτήτων για την επίλυση του προβλήματος του διεθνούς λοιμού και θα συνεχίσουμε να παίζουμε ενεργητικότατο ρόλο για να συνεισφέρουμε στη γενική τροφιμική ασφάλεια. Η έκθεση Μαγκίνες είναι μια πολύ καλή ανάλυση και θα μας δώσει ορισμένα κλειδιά που θα τα λάβουμε σοβαρά υπόψη μας και εμείς και οι διεθνείς κοινότητες. Ευχαριστούμε. Passamos ao relatório seguinte, que é Προχωρούμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Γενοβέφα Γκραμπόφσκα σχετικά με το διάλογο των πολιτών στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας. Τέσσερα λεπτά κυρία Γκραμπόφσκα. Μάικρο, please. I pressed. Thanks.